Κηρύττω την Σύνοδο του Κοινοβουλίου που διακόπη στις 20 Απριλίου 2012 ε, εκ νέου αρχίσασα. Τα πρακτικά της συνεδρίας 20 Απριλίου 2012 έχουν διανεμηθεί, υπάρχουν παρατηρήσεις ή αντίρρηση.